buongiorno colleghi la seduta è aperta Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, άρχισε η συνεδρίαση. Χθες ο πρόεδρος ανακοίνωσε μια ερμηνεία του άρθρου 166-167 παράγραφος 1 και 195 εδάφιο 3 του εσωτερικού κανονισμού. Πρόταση